Συνεχίζουμε με το σημείο υπαριθμών 5. Κατάλαβα ότι όλοι οι Ισπανοί έχουν αποχωρήσει. Ίσως έχει να κάνει κάτι με το ποδοσφαιρικό αγώνα. Η Γεωργία είναι πάντα στο μυαλό μου, όπως λέει και το αντίστοιχο τραγούδι. Ερχόμαστε στην έκθεση για τα θέματα προξενικών θεωρήσεων με τη Γεωργία. Η συγητής είναι ο κύριος Μαμικίνης. Η έκθεση επί της ουσίας είναι, γίνεται από την Μαρίγια Γκαμπριέλ. Και τώρα η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ προβλέπει να ψηφίσει την έκθεση της των ε, Σεπτέμβριο, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να επιταχύνουμε και εμείς και η πρότασή μας στις 21 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι να είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες και η ψηφοφορία θα γίνει στις 12 Ιουλίου. Γίνεται δεκτή αυτή η πρόταση. Εντάξει. Εντάξει, οπότε μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση στο, τη ψηφοφορία στο Στρασβούργο στις 7 Ιουλίου. Όσο πιο γρήγορα το κάνουμε, τόσο πιο πολύ μπορούμε να επηρεάσουμε τα τεκτενόμενα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Κύριε Μάμικη έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πρόταση της Κομισιόν είναι να τροποποιήσει τον κανονισμό 539 του 2010 ώστε να δοθεί ελευθερία από προξενικές ε, θεωρίες στους πολίτες γεωργίας που έχουν βιωματικά διαβατήρια. Η Συμφωνία για τις προξενικές θεωρίες και την επανεισδοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας ετέθησε εφαρμογή το Μάρτιο 2011. Η οριστική εφαρμογή αυτών των δύο συμφωνιών ήταν προαπαιτούμενο για την πρόθεση του διαλόγου για την φιλελευθερωποίηση προξενικών θεωρήσεων σε όλο αυτό το διάστημα η Κομισιόν εξέδωσε, εξέδωσε εκθέσεις προόδου σε σχέση με την, τα ζητήματα αυτά. Η τελευταία τέτοια έκθεση ενεκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2015 και η Κομισιόν εκεί συμπεραίνει ότι έχει γίνει απαραίτητη πρόοδος <clears throat> και όλα τα προαπαιτούμενα benchmarks έχουν επιτευχθεί. Η αυτή προφανώς θα ευνοήσει πολύ τους πολίτες της Γεωργίας, θα βοηθήσει τις επαφές μεταξύ πολιτών, απλών ανθρώπων, μεταξύ φοιτητών και επιχειρηματιών. Θα κάνει πιο ε, μεγάλη την ελκυστικότητα την γεωργία και για τους ε, ευρισκόμενους στην Αυχασία και την Οσετία, μειώνοντας τις ε, εντάσεις στις περιοχές αυτές. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνει το ταχύτερο δυνατό η ενέργειας για να εφαρμοστεί ο τροποποιημένο κανονισμό. Δεν κατανοούμε γιατί υπάρχει καθυστέρηση και χρονοτριβή στο Συμβούλιο, αλλά μόνο φήμε έχουμε από τα μέσα ενημέρωση, δεν έχουμε επίσημη πληροφόρηση και οι φήμε λένε ότι ο κύριο λόγο είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται με άλλε χώρε όπω η Ουκρανία, η Τουρκία και άλλες σημαντικές χώρες. Γιατί όμως να εξαρτάται από αυτές τις χώρες η αίτηση της γεωργίας και να τροχοπεδείται λόγω προβλημάτων με άλλες χώρες. Εγώ νομίζω ότι οι γεωργιανοί έχουν αλλάξει τους κανόνες στη χώρα τους, έχουν δεσμευτεί πάρα πολύ. Θα ήταν άδικο να μην προχωρήσουμε στη φιλελευθερωποίηση για τις προξενικές θεωρήσεις με τη Γεωργία. Η Γεωργία το περιμένει αυτό και η οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να θίξει τι σχέσει Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας, εξού και η σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα πρέπει να τονίσει ότι η Γεωργία κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσει να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατό το ελευθερία από προξενικέ θεωρήσει. Γι' αυτό η Επιτροπή μας θα πρέπει να ζητήσει από την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών που είναι η αρμόδια Επιτροπή να προτείνει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και έτσι να προχωρήσει σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στέτινα έχει το λόγο. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο είμαι σκιώδης εισηγητής και ασχολούμαι με τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Γεωργία οπότε και θα μπορώ παρά να επικρίνω αυτές τις προσπάθειες που γίνονται όσον αφορά την απελευθέρωση του καθεστώτου διαθέωσης διαβατήριων. Έχουμε επίσης και τη Συμφωνία Σύνδεσης που υποχρεώνει την χώρα να μπορέσει να ε, αναδεχθεί ε, αυτά τα ε, πρότυπα και το κεκτημένο στον πρώτο κράτος δικαίου, τα δικαιώματα και μιλούσαμε για τη λειτουργία τη αντιπολίτευση και είπαμε ότι είναι πάρα πολύ απαραίτητο να υπάρχει μια αντιπολίτευση, ούτω ώστε να είναι υγεία στο πολιτικό σύστημα. Και η αδίποτε πράξη ε, βία, οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά πολιτικού κόμματο θα πρέπει να ερευνάται αμελητή. Επίση, είπαμε ότι είναι απαραίτητο το ότι πάρα πολλοί από την αντιπολίτευση ακόμα βρίσκονται φυλακισμένοι. Και έχω επίσης αναφερθεί στο ότι ασκείται πολιτική πίεση ε, και ε, επίσης η κυβέρνηση επηρεάζει την δικαιοσύνη αλλά και την ελευθερία έκφρασης. Εν κατακλείδη για την ε, Γεωργία θα πρέπει να πούμε ότι διατρούν πάρα πολλέ επιφυλάξεις. Το πολιτικό τοπίο της χώρας πολλώνεται όλο ένα και περισσότερο ακριβώς επειδή σύντομα θα γίνουν εκλογές, επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης. Ε, αυτές οι επιθέσεις δεν ερευνούνται από τη δικαιοσύνη ή ερευνούνται με στοιχειώδη τρόπο, έχουμε κάποια σκάνδαλα, έχουμε ε, κάποιες ε, καταδίκες στελεχών του Υπουργείου Αμήνης ε, σε κάποιες δίκες που δεν είναι καθόλου δίκες. Επίσης έχουμε καταγγελίες από την Ένωση Νέων Δικηγόρων. Ισχυρίζονται ότι οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση αυτή ήταν αθώοι. Πάντως αύριο περιμένουμε την ε, απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, για την περίπτωση κυρίου Βίσου Ασφίλη. Και Θέλουμε να δούμε τι θα γίνει, κατά πόσο θα μπορέσει αυτή η χώρα να πλήρει τι προποθέσει που έχουν ταχθεί και η ευελιξία που έχουμε δείξει να μην θεωρηθεί αδυναμία και επιταγή είναι λευκό. Κύριε Μάμπικινς, αν μπορέσετε στην ε, αιτιολογική σας ε, έκθεση να αναφέρετε αν μπορέσετε αυτά τα οποία σα είπα. Ο πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Thank you, Chair. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και συμφωνώ με όλα όσο είπε ο κύριο Στέτινα. Έχουμε υπόψη μας ε, όλα αυτά τα οποία γίνονται στην χώρα και το τι επικρατεί όσον αφορά την επίθεση στην αντιπολίτευση. Θα πρέπει επομένως να δούμε και το πολιτικό τοπίο της χώρας διότι φοβούμε πως η αδίποτε αναβολή και δισταγμός όσον αφορά το θέμα των θεωρήσεων διαβατηρίου θα είναι κάτι πολύ αντιπαραγωγικό. Άρα θα πρέπει να ζυγίσουμε τα πράγματα με μεγάλη προσοχή. Όλα τα βασικά πολιτικά φιλοδυτικά κόμματα ομονοούν για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα τέτοιο ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση της χώρας. Το ότι θα πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης. να βρεθεί μια λύση στο θέμα των ε, φυλακισμένων στελεχών της αντιπολίτευσης. Και φυσικά θα είναι αντίστοιχη με αυτά που λέμε εμείς, ελπίζουμε η απόφαση του Δικαστήριου του Στασβού για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Πολύ σημαντικό όλα αυτά δεδομένες της σημερινής πολιτικής συγκυρίας. Ελπίζουμε τα πράγματα να πάρουν μια καλύτερη ρότα και με τη βοήθεια της ε, θετικής απόφασης του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο δίνει τον λόγο στον κύριο Αστραβίτσιος. Η Γεωργία έχει υπογράψει τη Συμφωνία Σύνθεσης και είναι έτοιμη να την εφαρμόσει. Και δεν πρόκειται ε, μόνο για ελεύθερο εμπορίου συμφωνία, πρόκειται για ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών. Εμείς σεβόμαστε ακόμα τη συμφωνία αυτή και πρέπει να ολοκληρωθεί με την υλοποίηση. Και άπαξ και η Γεωργία κάνει αυτά τα οποία περιμένουμε από αυτή να κάνει, να εφαρμόσει δηλαδή όλες τις διατάξεις όσον αφορά την κατάργηση της θεώρησης, τότε θα πρέπει και εμείς να είμαστε ειλικρινεί και να πάρουμε την απόφασή μας. Ξέρω ότι μερικές χώρες βλέπουν ακόμα λόγους για καθυστέρηση, αλλά εγώ πιστεύω ότι τη συμφωνία αυτή πρέπει να την προχωρήσουμε αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς σωστοί εταίροι. Όντως, πολλά είναι τα ζητήματα ο συνάδελφος Τέτιν έχει δίκιο. Πρέπει να ελέγξουμε την κατάσταση. Πρέπει να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι για όλα τα σημεία, για τη δημοκρατική διαδικασία και τον έλεγχο κυρίως, αλλά η κατάργηση της θεώρησης είναι μια πολύ σημαντική απόφαση που περιμένουν οι Γεωργιανοί πώς και πώς. Η Επιτροπή μας λοιπόν θα έπρεπε να αποφανθεί θετικά και έγκαιρα με μια λύση προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο λαός της Γεωργίας. Και πιστεύω ότι το αξίζουμε απόλυτα. Αξίζει να ζουν σε ένα κράτος το οποίο συνάδει με όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό σημαίνει όχι επιλεκτική δικαιοσύνη, όχι πολιτική κρατούμενη, ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής και ελεύθερες εκλογές. Θα πρέπει να σταματήσει να παρενοχλεί τις απαραίτητες ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης η Γεωργία, όπως το Ρουστάβι και να είναι μεροληπτική στο διορισμό των μελών του ανώτατου δικαστηρίου. Εξακολουθούν να είναι ε, αντιπολιτευόμενοι, η προηγούμενη κυβέρνηση ουσιαστικά, στη φυλακή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αλλά παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να καθυστερήσει την ε, χορήγηση ελευθερία από προξενικέ θεωρήσει, αλλά και να θεσπίσει ένα φρένο ασφαλεία εάν η Γεωργία δεν τηρήσει τα ευρωπαϊκά δημοκρατικά πρότυπα. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρο. Νομίζω η Κομισιόν θα μπορεί να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα, εφόσον το, το επιθυμεί βέβαια, γιατί ένα από τα ερωτήματα έχει να κάνει με το λεγόμενο φρένο ασφαλείας για τα θέματα αυτά. Φυσικά θα πρέπει να εγκριθεί πρώτα μια τέτοια δικασία, ώστε στη συνέχεια για ορισμένα μπορούν να αρθούν οι αντιρρήσεις τους, ώστε να προχωρήσουμε στη φιλελευθερωποίηση προξενικών ε, θεωρήσεων. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν θα ήθελε να λάβει το λόγο για το θέμα αυτό. Εάν λοιπόν υπάρξει, υπάρχουν, ε, εάν δεν υπάρξει μια τέτοια ρύθμιση, κάποιες χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία μπορεί να εμποδίσουν την ε, απόφαση για λόγους ε, ασφαλείας. Και υπάρχουν και εκπρόσωποι των γεωργιανών συμμοριών, όχι τραπεζών λέει ο πρόεδρος, με διορθώντας το σαρδάμ του, οι οποίοι δημιουργούν κάποιες ανησυχίες σε μας. Εν Υπάρχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή ως πολιτικοί κρατούμενοι και είναι απαραίτητο να ε, απελευθερωθούν κατά την άποψη πολλών βουλευτών και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί και είναι ένα θέμα που αφορά και την εσωτερική ασφάλεια στα πλαίσια της ε, γεωργίας. Ποια είναι η θέση λοιπόν, ποια είναι η άποψη της Κομισιόν για να μην δημιουργηθεί και πρόβλημα για την εσωτερική ασφαλεία, ασφάλεια των πολιτών της Ευρώπης λόγω της προξενικής αυτής αφελευθέρωσης. Σας ευχαριστώ, λέω εκπρόσωπος της Κομισιόν. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του προς την πρόταση της Κομισιόν, κάτι το οποίο χαιρετήσουμε. Προσβλέπουμε επίσης να μπορέσει να ευδοκιμήσει αυτό το θέμα και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για το ερώτημα το οποίο έθεσε ο πρόεδρος για τη σύνδεση με το μηχανισμό φρένου ασφαλείας του μηχανισμού αναστολής. Στις 4 Μαΐου έκανε μια πρόταση για τη θέσπιση του μηχανισμού αναστολής Κομισιόν και χαιρόμαστε για το γεγονό ότι το Κοινοβούλιο θα διεκπαιρεώσει το θέμα αυτό το ταχύτερο δυνατό. Το, το Συμβούλιο στις 20 Μαΐου συμφώνησε για μια γενική προσέγγιση και τώρα εναπόκειται για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ με τον κύριο Μέρα να παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσή του στην Επιτροπή Λίμπερ. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει αύριο. Υπάρχει η απαραίτητη σπουδή λοιπόν και πιστεύω ότι όλες οι ανησυχίες για το θέμα αυτό θα μπορέσουν να ξεπεραστούν. Για το οργανωμένο έγκλημα δεν γνωρίζω ακριβώς σε τι αναφέρεται ο πρόεδρος αλλά εμείς στο βαθμό που γνωρίζουμε ξέρουμε ότι αυτό έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο αλλά τα benchmarks για το οργανωμένο έγκλημα από την πλευρά της Γεωργίας έχουν εκπληρωθεί. Για το πιο συγκεκριμένο θέμα που εγείρει ο πρόεδρος δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Πότε προβλέπετε λοιπόν να αποφασιστεί το, η διαδικασία αναστολής το φρένο ασφαλείας στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο για τη χρονική αλληλουχία των πραγμάτων. Ο μηχανισμός αυτός ε, αναστολής, το φρένο ασφαλείας που λέτε, υπάρχει ήδη μια συμπεφωνημένη γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο που ενεκρίθη στις 20 Μαΐου και στο Κοινοβούλιο, όπως γνωρίζετε, εναπόκειται στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ με εισηγητή τον κύριο Θεμέρα και από ό,τι καταλαβαίνουμε θα παρουσιαστεί η έκθεσή του αύριο στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Την ε, Τετάρτη μάλλον, την Τετάρτη αυτής της εβδομάδας. Και θεωρούμε ότι πριν από τις θερινές διακοπές θα υπάρχει, θα γίνει ψηφοφορία η 12 ή 13 Ιουλίου στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Αν γίνει λοιπόν κάτι τέτοιο, αν επιτευχθεί αυτό στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ λέτε, τότε θα έρθει στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο, λέει ο πρόεδρος. Οπότε μπορεί να γίνει το άλλο πράγμα τον Οκτώβριο, λέει ο κύριος Μπλοκ. Αλλά πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στο χρονοδιαγράμμα else? Η Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να προσθέσω ότι στην πρόσφατη επίσκεψη της ΕΝΤΕ στη Γεωργία, της Υποπιτροπής ε, δηλαδή, συζητήσαμε με τον Υπουργό Εσωτερικών εκεί και εκείνο μας ενημέρωσε επιμακρό για τις προσπάθειες που κάνει το Υπουργείο του αλλά και οι λοιπές αρχές της Γεωργίας προκειμένου να συνεργαστούν με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προκειμένου να μπορέσουν να καταπολεμήσουν κάθε δράση συμμοριών. Νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς να δούμε λίγο τις στατιστικές των χωρών μελών και η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια είναι πάρα πολύ δύσκολη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πολλούς και διάφορους λόγους βέβαια. Οι γεωργιανοί πολίτες που προχωρούν σε εγκλήματα δεν είναι οι περισσότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε προσοχή. Ελπίζω να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Εντάξει, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση σε μια μεταγενέστερη ευκαιρία. Και φυσικά θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο αυτό της φιλελευθερωπής το ταχύτερο δυνατό προς το συμφέρον της γεωργίας, χωρίς βέβαια να δημιουργηθεί εντύπωση ότι υπάρχει ανασφάλεια, ότι θα δημιουργηθεί ανασφάλεια μεταξύ των πολιτών μας λόγω αυτής της ρύθμισης και δεν θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα σε κάποιους να την εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Θα πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι και εναντί του πληθυσμού μας με την συμφωνία αυτή. κύριε Σιγητά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Ευχαριστώ για όλες αυτές τις απόψεις που μεταφέρατε εδώ. Ως εισηγητής θα λάβω υπόψη μου τις παρατηρήσεις σας. Και από τη δικιά μου την πλευρά το μόνο που έχω να προσθέσω και να επαναλάβω είναι τα λόγια ε, ημών κυρία Μπρόκ στο Στρασβούργο που είπατε ότι η κατάργηση θεωρήσεων είναι ένα δώρο προς τον πληθυσμό της Γεωργίας, προς τους πολίτες τους, ένα δώρο που χρειάζονται. Όλες ε, οι χώρες που έχουν περάσει από κατοχή το χρειάζονται αυτό. Σίγουρα θα το εκτιμήσουν όλος ιδιαίτερος οι Γεωργιανοί. Τώρα οι συμμορίες και ό,τι άλλα παράνομα πράγματα γίνονται, εννοείται ότι δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Πάντως να ξέρουμε ότι το θέμα τη κατάργηση τη θεώρηση είναι πολύ σημαντικό για τον λαό εκεί, για του ίδιου του Γεωργιανούς. Χωρίς μικρόφωνο ο πρόεδρο. Έχουμε το επόμενο σημείο στις 16.45. Μπορούμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Meine Damen und Herren. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Συγγνώμη γιατί δεν είναι πολύ μεγάλη η προσέλευση, αλλά είναι πολλοί βουλευτές που είναι με την ε, συνάντηση των ΑΚΕ στην Ναμίμπια, η οποία έχει μεγαλύτερη γοητεία από τις Βρυξέλλες ίσως και κλιματολογικά. Αλλά υπάρχουν πολλοί που μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο μέσω web streaming. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω ιδιαίτερα εγκάρδια κύριε Κρέεν Μπιουλ για το γεγονός ότι είσαστε διαθέσιμος να μας παρουσιάσετε την ε, κατάσταση σε σχέση με τους Παλαιστίνους πρόσφυγες και την ε, παροχή χρηματοδοτικών μέσων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό το έργο σας. Θα θέλαμε λοιπόν την ε, άποψή σας σε σχέση με την κατάσταση στη Γάζα mm. και την άποψή σας σε σχέση με τις πρόσφατες εξέλιξεις που έχουν λάβει η χώρα μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω το λόγο να του παρουσιάσετε τα θέματα αυτά στα μέλη της Επιτροπής μας. Παρακαλώ, ναι. Και στο τέλος θα μπορούσε να λάβει το λόγο και ο εκπρόσωπος της ε, Κομισιόν, κ. Βάβενη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά είμαι και πάλι ενώπιόν σας πρόσκληση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχω την ε, ευκαιρία να παρουσιάσω ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου το έργο της ε, Ούνορα σε μια πολύ δύσκολη και ασταθή Μέση Ανατολή. Η παρουσίαση αυτή βέβαια λαμβάνει χώρα σε μια πάρα πολύ ταραγμένη εποχή στη Μέση Ανατολή, σε μια χρονική στιγμή όταν η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα αποτελέσματα της αστάθειας στη Μέση Ανατολή, τις εντάσεις, τις προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τον αριθμό των προσφύγων, τον μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων που έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχρόνως βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η UNRWA θέλει να υπογραμμίσει την κατάσταση και τα βάσανα των Παλαιστινίων προσφύγων στο ευρύτερο πλαίσιο της ε, Μέσης Ανατολής και τις σημαντικές προσπάθειες που έχει καταβάλει η UNRWA για να ανακουφίσει τα προβλήματά τους. Και <clears throat> φυσικά θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κάτι μέλη της για την ιδιαίτερα γενναιόδορη υποστήριξη που έχουν δώσει προς την UNRWA στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων της. Έχουν περάσει πια 45 χρόνια από τη χρονική στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε τη διαρθρωμένη υποστήριξή της προς την Ούνρα. Και άμα σκεφτείτε ότι η Ούρα βρίσκεται σε λειτουργία μόνο 65 χρόνια, αυτό είναι φόρος τιμής στην ε, στεναρότητα, την προβλεψιμότητα και την ποιότητα της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ούνρα. Θέλω ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου προς το Κοινοβούλιο και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μόνιμο ενδιαφέρον τους και τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους στο θέμα των Παλαιστινίων προσφύγων και της Σούντζα. Θέλω ευχαριστήσω και την Κομισιόν και το Συμβούλιο για τον, την υποστήριξη του έργου της ΣΟΥΡΑ και τη συμβολή που κάνουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Μέσης Ανατολής. Είσαστε <clears throat> από κοινού οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τα κρατη η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης προς την Ούντρα, κάτι το οποίο φυσικά μας κάνει να είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες. Θα ήθελα να ξεκινήσω υπογραμμίζοντα μια σειρά θεμάτων που έχουν να κάνουν με το γενικό πλαίσιο στο οποίο εργάζεται η Ούνδρα. Όπως ξέρετε, είμαστε ένα φορέα που έχει ως εντολή εδώ και 66 χρόνια να δραστηριοποιηθεί στην ε, Δυτική Όχθη, τη Γάζα, τη Σύρια, την ε, Συρία, η Ορδανία και Λίβανο. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες σε αυτές τις χώρες. Και στη συνέχεια μπορώ να σταθώ σε κάποιες από τις επιτυχίες της ώρα το ρόλο μας και τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν σας και να σας εκφράσω επίση και κάποιες σκέψεις για το πού θα ήταν πολύ σημαντικός ο ευρωπαϊκός ρόλος στις επερχόμενες εβδομάδες και μήνες. <clears throat> Από πολλές απόψεις η κατάσταση των Παλαιστινίων προσφύγων στη Μέση Ανατολή είναι μια κρίση υπαρξιακή για τους πρόσφυγες αυτούς ουσιαστικά. Ένας από τους λόγους αυτής της κατάστασης είναι ότι η προσοχή της κοινή γνώμης, της διεθνούς κοινή γνώμης για την κατάσταση των Παλαιστινίων προσφύγων έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το κατανοούμε φυσικά ενώπιον της μεγάλης καταστροφής που βλέπουμε στη Συρία, το Ιράκ και την Ιεμένη, την προσοχή που έχει στραφεί προς την Λιβύη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δικαιολογημένα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε 5,2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες που ζουν στη Μέση Ανατολή σε πολύ ασταθείς συνθήκες και δεν πρέπει η παγκόσμια κοινή γνώμη να παραγνωρίσει αυτό το πρόβλημα. Ένα παράδειγμα είναι αυτό το οποίο είδατε να συμβαίνει στη Δυτική Οχθή τους τελευταίους μήνες. Ξέρουμε ότι η Δυτική Οχθή και η Ανατολική Ιερουσαλήμ γνώρισαν μια ανασωπήρωση δράσεων βίας και διαδηλώσεων υπήρξαν πράξεις βίας που έπληξαν άμαχους, Παλαιστινίους αλλά και Ισραηλινούς σε αυτό το χρονικό διάστημα. Όλα αυτά καταδεικνύουν πόσο μεγάλη απόγνωση υπάρχει πια στα κατεχόμενα εδάφη της Παλαιστίνης και πρέπει να θυμόμαστε ότι του χρόνου θα φτάσουμε 50 χρόνια κατοχής της Δυτικής Όχθης και της Γάζας. Είναι ουσιαστικά όλη η δική μου πορεία στη ζωή. Από τη στιγμή που γεννήθηκα, αν είχα γεννηθεί στην Ευρώνα, στην Τζενίν ή κάπου στη Γάζα, θα είχα ζήσει τα 50 χρόνια της ζωής μου κάτω από κατοχή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μην το ξεχάσουμε γιατί έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις για τους πολίτες εκεί. Όταν επεκτείνονται οι επικισμοί, όταν ανατινάσσονται τα σπίτια των Παλαιστινίων, όταν υπάρχουν κίνδυνοι να μεταφερθούν σε άλλες περιοχές και όταν περιορίζονται οι προοπτικές για τα άτομα αυτά, αυτό φυσικά τροφοδοτεί την αστάθεια. Όλα αυτά τα οποία έχετε δει στο χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2015 με την αυξανόμενη ε, αναταραχή στα Παλαιστινιακά εδάφη, όλο αυτό προέρχεται από νέους που έχουν γεννηθεί μετά από την Συμφωνία του Όσλο, που τους έχουν πει ότι αν πιστέψουν στην πολιτική διαδικασία, αν είναι μετριοπαθείς στην πολιτική τους δράση, θα υπάρξει μια αμοιβή. Δεν έχουν δει καμία τέτοια αμοιβή. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν με προσδοκίες οι οποίες έχουν ματαιωθεί απόλυτα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα πάψουν, είναι φυσιολογικό να πάβουν να πιστεύουν ότι η πολιτική δράση μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Στη λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή το σορευτικό αποτέλεσμα πιέσεων και περιορισμών για, τους, ε, για τον πληθυσμό της Γάζας που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για το μέλλον της Λόριδας της Γάζας. Πρέπει να το τονίσω αυτό από την οπτική γωνία ενός φορέα ο οποίος εργάζεται ιδιαίτερα στη Γάζα. 70% από τα 1,8 εκατομμύρια των ε, πολιτών της Γάζας είναι Παλαιστινοί πρόσφυγες. Επομένως η ώρα έχει άμεση ευθύνη για να τους παρέχει βασικές υπηρεσίες, παιδεία, υγειονομική περιθέλψη κτλ. Στη λωρίδα της Γάζας με ρωτάνε πολλές φορές πόσο έχουμε προχωρήσει για την ανοικοδόμηση. Έχει προχωρήσει η ανοικοδόμηση στη Γάζα, όχι αρκετά γρήγορα, όχι ικανοποιητικά για όλους αυτούς που χάσαν τις οικίες τους και τις αιστείες τους στον πόλεμο του 2014. Κάτι όμως το οποίο με ανησυχεί πολύ περισσότερο από την καταστροφή των κτηρίων και των υποδομών είναι το εξή. Μπορείτε να φωτογραφίσετε ορισμένε περιοχέ τη Γάζα πριν από το 2014 και να δείτε ποιο ήταν το επίπεδο καταστροφή που έλαβε χώρα στον πόνο του 2014. Μπορείτε σήμερα να φωτογραφίσετε πάλι αυτή την περιοχή και να δείτε το επίπεδο της καταστροφής με το επίπεδο της ανοικοδόμησης. Αυτό όμως που δεν μπορείτε να δείτε είναι να καταγράψετε τον ψυχολογικό αντίκτυπο που έλαβε χώρα στους ε, ζώντες στην Γάζα. Αυξάνονται οι αυτοκτονίες στην λόγια της Γάζας, που στο παρελθόν ήταν πάρα πολύ μικρό το ποσοστό αυτοκτονιών, γιατί ο ίδιος ο κοινωνικός ιστός, οι κοινότητες των πολιτών της Γάζας έχουν διαραγεί, γιατί δεν υπάρχουν προοπτικές. 90% από τα 250.000 παιδιά Παλαιστινίων που πηγαίνουν σε σχολεία τη Σούρα στη Γάζα δεν έχουν βγει ούτε μια φορά στη ζωή του από τη λωρίδα τη γάζα. 90% από αυτά τα παιδιά. Και οι υπολογισμοί μα, επί τη βάση των στοιχείων που έχουμε για το 2015, μόνο 10.000 άτομα έφυγαν πέρσι από τη λωρίδα τη Γάζας. Αν τα 1,8 εκατομμύρια ατόμων που ζουν στην περιοχή τη Γάζας μπουν σε αυτόν τον υπολογισμό, Μόνο κάθε 180-200 χρόνια έχει κάνει την ελπίδα να φύγει από τη, από τη Γάζα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και αυτοί που παίρνουν από τα σχολεία μα και έχουν περάσει 9 χρόνια παιδεία βγαίνουν με προσόντα, με κίνητρα, με ενθουσιασμό για να συμβάλλουν στην κοινωνία του, αλλά δεν θα βρουν ποτέ μια δουλειά οι περισσότεροι από αυτού. 65% των νέων Παλαιστινίων στη Λωρίδα τη Γάζα είναι χωρί εργασία. 65% αν αυτό δεν είναι το υψηλότερο ποσοστό ανεργία στον κόσμο, είναι από τα υψηλότερα. Πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν μπορώ να δω πώς εν ώψη αυτών των παραμέτρων μπορούν αυτά να συνάδουν με την εξασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή, όσο θεμητές και να είναι αυτές οι ανησυχίες για ασφάλεια. Δεν μπορεί κανείς να έχει ασφάλεια και σταθερότητα σε μια περιοχή που 65% των νέων είναι άνεργοι. Παρά το γεγονός ότι έχουν κατάρτιση και εκπαίδευση και δεν μπορούν να φύγουν από τη Γάζα. Το μόνο που μπορεί να υπάρξει είναι να αισθάνονται απογοήτευση ε, και ματίωση. Οπότε αυτά θα πρέπει να σκεφτεί όταν προβληματίζει για τη Γάζα και επίση να σα αναφέρω ότι ένα από του μεγαλύτερου κινδύνου που έχουμε όποτε προσπαθούμε να τα αναλύσουμε τα πράγματα από πλευρά ανθρωπιστική αλλά και πλευρά είναι το ότι θέλουμε ε, τελικά να μην βλέπουμε ανθρώπου αλλά νούμερα και στατιστικά. Όμως θα πρέπει να το δούμε ανάποδα πράγματα. Πριν από λίγες μέρες, ξέρετε, είχαμε έναν δάσκαλο που πήγε εκεί και αυτή η κοπέλα ε, οργάνωσε έναν διαγωνισμό με θέμα τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ήταν πολύ απογοητευμένη από γιατί από ό,τι μου είπε αυτός ο διαγωνισμός στο σχολείο της απέτυχε. Τι ρωτώ γιατί. Γιατί κανένας από τους μαθητές δεν μπόρεσε να προτάξει, να προβάλλει ένα όραμα, ένα όνειρο. Βλέπετε αυτό συμβολικά πόσο, πόσο νόημα έχει, ε, τι, τι, τι αισθάνονται εκεί ο κόσμος για το αν μπορεί να μετακινηθεί όχι. Και έχουμε επίσης την κατοχή της Δυτικής Όχθης ε, και αν πάει κανείς στην Συρία, πριν από ένα μήνα πήγε τελευταία φορά και είδα εγώ διάφορες καταστάσεις που με ε, συνετάραξαν πολύ και πέραν του, του ευρύτερου της τραγωδίας του πολέμου έχουμε και μια τραγωδία που αφορά ε, Παλαιστίνους πρόσφυγες. Πριν από τον πόλεμο ήταν εκεί 5.600 και παραμένουν ακόμη πρόσφυγες 120.000 έχουν φύγει από τη χώρα και η μισή πήγαν σε Ιορδανία και Λίβανο. Άλλοι από αυτούς τους πρόσφυγες πήγαν στην Τουρκία ή την Αίγυπτο. Και πολλοί από αυτούς μπόρεσαν να φτάσουν στην ε, Ευρώπη κυρίως από το καλοκαίρι και μετά. Και αυτό το που γίνεται είναι ότι φεύγουν από διάφορες τοποθεσίες που έχουν καταστραφεί τώρα, ε, είχαν στατόπεδα και τώρα φτάνουν στην πρώτη γραμμή του πυρός, καταστροφές ε, και από βομβαρδισμούς και από πυροβολικό, από κάποιους βομβιστές καμικάζι ε, και μέσα στη Δαμασκό γίνανε αυτά ε, και εκεί σε μια γειτονιά Παλαιστινίων είχαμε επιθέσεις που τους χτύπησαν, οπότε θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι στην Σύρια ε, πάντοτε ήταν καλοδεχούμενοι οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες δουλειές, είχαν μαγαζιά, επιχειρήσεις στέλνανε στα σχολεία μας τα παιδιά και θεωρούσαν ότι έχουμε καλό επίπεδο παιδείας, αλλά χρειαζόταν την γόνορα για άλλες δραστηριότητες. Είχαν τέλο πάντων μεγάλη αυτάρκεια για να καλύψουν την οικογένειά τους. Τώρα το 90% αυτών ε, εξαρτώνται τελείως από τη δική μας υπηρεσία. Και η νέα γενιά αισθάνεται ότι είναι βέβαια μια ανάμνηση τραγωδία του 48 και ας αναφέρονται σε αυτή ακόμα γονείς και παπούδες, αλλά δεν έχουν άμεση παράσταση. Τώρα με αυτό που ζουν καταλαβαίνουν τι πέρασαν οι παππούδες και οι γονείς. Άλλη γενιά Παλαιστινίων τώρα και όμως αυτοί τώρα στο πετσί τους βλέπουν τι θα πει απώλεια, ε, τι θα πει απώλεια οικογένειας, ε, γειτόνων, ε, και βλέπετε ποιο είναι το τοπίο όσον αφορά τους Παλαιστινίους πρόσφυγες στην Μέση Ανατολή. Έχουμε 5,2 εκατομμύρια οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν σε αυτό το μεσανατολικό τοπίο που χαρακτηρίζεται από τόση αστάθεια με όλους αυτούς τους πολέμους, συγκρούσεις που γνωρίζουμε. Να, ακόμα ένας παράγον κινδύνου για την περιοχή, εάν δεν κάνουμε κάτι για το τι χρειάζονται, γιατί να τους δώσουμε την αξιοπρέπειά τους και να το κάνουμε και δυναμικά. Και υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, το ότι δεν υπάρχει κάποιο πολιτικό όραμα για αυτούς. Η ούνρα δεν είναι πολιτική πλατφόρμα, δεν έχουμε έντολη για πολιτικό έργο, αλλά καθημερινά αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι σε ανθρώπινο επίπεδο τι πάει να πει έλλειψη πολιτικού ορίζοντα. Δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα για να γίνουν κάποιες πολιτικές εξελίξεις όσον αφορά το Παλαιστινιακό, την αντιπαράσταση με, την, με το Ισραήλ, αλλά επίση και το πρόβλημα όσον αφορά την Συρία. Και πρόκειται για πολύ σημαντικά ζητήματα, αν είναι οι Παλαιστίνοι δεν μπορούν να φανταστούν μια επιστροφή σε μια διαδικασία όπου μπαίνουν αυτοί στο προσκήνιο και ότι υπάρχουν προοπτικές ε, πρόοδου και τότε το πρόβλημα μόνο θα φουσκώνει, θα μεγαλώνει. Και ακριβώς ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτό, η έλλειψη του πολιτικού ορίζοντα. Τώρα, για να στραφούμε στις τη της Ούνρα ε, ε, για να δείτε πού στιάζουν προσοχή μας, να δείτε και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Όπως προείπα, επί 65 χρόνια έχουμε αναλάβει δράση στην περιοχή, σε κάποια ε, σημεία κλειδιά και όταν εγώ μπήκα στην υπηρεσία ε, ήταν για μένα μια αποκάλυψη. Η πρώτη εμπειρία μου που είναι σημαντικό να σας την πω είναι το τι γίνεται με την παιδεία, την εκπαίδευση η επένδυση που κάνουμε και που εσείς ως Ευρωπαίοι, εσείς ως βασικοί εταίροι αυτής της προσπάθειας είναι το πώς θα εκπαιδεύσουμε αυτούς τους νέους Παλαιστινίους. Ό,τι πιο σημαντικό έχει γίνει ποτέ στη Μέση Ανατολή σε επίπεδο ανθρωπιστικό και θα πρέπει επομένω να αναγνωρίζουμε, να γνωρίζουμε περισσότερο τους εταίρους και τους δωρητές. Πάνω από 500.000 αγόρια και κορίτσια από την Παλαιστίνη ε, φοιτούν στα σχολεία μας. Μιλάμε για 700 σχολεία στη Μέση Ανατολή. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το συγκρίνουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Βέβαια, Νέα Υόρκη και ο Λος Άντζελες είναι τα πιο μεγάλα <clears throat> εκπαιδευτικά δίκτυα, αλλά καθίστε και συγκρίνετε αυτά τα 700 σχολεία σε σχέση με το τι γίνεται στην Ευρώπη και μάλιστα μέσα σε ένα τοπίο πολέμου και την Είπαμε για 5,2 εκατομμύρια προσφύγων. Οπότε αυτά τα αριθμητικά στοιχεία δεν είναι τόσο γνωστά. Όμως μιλούμε για 40% των μακροχρονίων προσφύγων όλου του κόσμου είναι αυτό το, αυτό το σαν αυτή η Παλαιστίνη. Και αυτό σας λέω ότι η Ούνορα, η υπηρεσία μας, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο με το που βοηθά αυτή την κοινότητα. Μιλάμε για 500.000 μαθητές, 3 εκατομμύρια ασθενείς τα νοσοκομεία μας και 1,5 εκατομμύριο που ωφελούνται από αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια. Πρόκειται για μια συμβολή στη σταθερότητα της περιοχής και στην στήριξη της αξιοπρέπειας του κόσμου αυτού. Πολλές φορές υποτιμάται το τι θα συνέβαινε εάν η Ούνρα δεν μπορούσε να παρέχει αυτές τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Ξέρετε, ένα χρόνο πριν, λίγο μετά την επίσκεψη που έκανε στην Επιτροπή σας, αντιμετωπίσαμε το μεγαλύτερο οικονομικό μας πρόβλημα στην ιστορία μας. Μας λείπανε 100 εκατομμύρια δολάρια και θα έπρεπε γι' αυτό το λόγο να αναβάλουμε την έναρξη του σχολικού έτους. Για όλα αυτά τα 700 σχολεία καταλαβαίνω ότι νιώθετε πάνω Δηλαδή έχω τρία παιδιά. Φανταστείτε τι πάνω να τους πω των παιδιών μου, των αγοριών μου ότι αναβάλλεται για κάτι εβδομάδες, για κάτι μήνες του σχολείο. Θα πανηγυρίσουν, αλλά στην περιοχή αυτή ήταν τραγωδία, γιατί εκεί η παιδεία θεωρείται το, το, το στήριγμα, η σημαία της ταυτότητάς τους, τη αξιοπρέπειά τους. Και ακριβώς η παιδεία να βρίσκεται εν κινδύνο ήταν ένα σοκ για όλη την κοινότητα. Είναι κάτι που συντάραξε όλες τις χώρες της περιοχής. Και ο Πρωθυπουργός της Ιορδανίας ε, ανέλαβε πολύ σημαντική πρωτοβουλία, προσπάθησε να βοηθήσει γι' αυτό τα 100 εκατομμύρια δολάρια που λείπανε, αλλά και ο Πρωθυπουργό του Λιβάνου τους Παλαιστινίους ηγέτες επίσης και άλλες χώρες και το Ισραήλ επίσης βοήθησε για να μπορέσουν να ανοίξουν τα σχολεία στην ώρα τους. Και δεν ήταν μόνο το δικαίωμα στην εκπαίδευση, ήταν το ότι οι 500.000 των Παλαιστινίων θα βρισκόντουσαν στον δρόμο εκτό σχολείων μεσούσε τη εκπαιδευτικής περίοδου. Ε, αυτό είναι το, το, πιο επικίνδυνο που μπορεί να γίνει. Και γι' αυτό σα λέω ότι η UNRWA είναι σημαντική και ότι η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει την ε, UNRWA. Ε, πρόκειται για μια επένδυση όχι μόνο Ισόφελος τη της αξιοπρέπεια, αλλά και ισόφελος τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτό να λάβετε υπόψη. Άλλες παράμετροι τώρα που αξίζει να αναφέρουμε όταν μιλούμε για τη βοήθεια σα προ την Ούλρα θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι είμαστε μια υπηρεσία που άμεσα δίνει αυτή τη βοήθεια με αυτή την ανθρωπιστική αερογή. Έχουμε όλο και περισσότερες υπηρεσίες και περισσότερο κόσμο που υλοποιεί αυτά τα οποία κάνουμε. Άρα βοηθάται οικονομικά μια υπηρεσία που αυτή την υπηρεσία ε, την μετακυλεί στους ε, εταίρους μας και φυσικά αυτό γίνεται με διοικητικές δαπάνες που καταβάλουμε. Επομένως η είναι το σημείο εισόδου και το σημείο εξόδου για ε, αυτή την βοήθεια και σας το λέω με, με, με τριοφροσύνη και με περηφάνεια ότι 98% του προσωπικού που βοηθάει είναι Παλαιστίνοι. Και συμμετέχουν παντού, στην πρώτη γραμμή, από το Χαλέπι, στο Χανιούνις, σε τόσες προβληματικές ε, περιοχές και πόλεις, για να υλοποιήσουμε, για να αναπτύξουμε τις δραστηριότητε παντού. Μιλάμε για 22.000 προσωπικό ε, νοσοκόμους, γιατρούς, δάσκαλους. Άρα τα λεφτά πιάνουν τόπο στην ούνρα γιατί φτάνουν στην κοινότητα. Πάμε στις υπηρεσίες υπέρ των Παλαιστινίων, αλλά είναι και η μισθή ε, των Παλαιστινίων υπέρ της κοινότητάς τους. Και είχαμε εκείνη σαν τις κορυφής για την ανθρωπιστική αρρωγή και είπαμε το πώς θα συνδυάσουμε, θα συγκεράσουμε ανθρωπιστική αρρωγή και ανάπτυξη. Πώς αυτές οι δύο δραστηριότητες λοιπόν θα συνδυαστούν όσο γίνεται καλύτερα και πριν από 65 χρόνια αυτοί που ίδρυσαν την UNRWA σκέφτηκαν το ότι είναι φυσικό να συνδυαστούν αυτές οι δύο δραστηριότητες στη ΔΕ Γάζα κατά τον πόλεμο ανοίξαμε 90 σχολεία και εκεί εφήλισαν 300.000 εκτοπισμένοι και οι δάσκαλοι τελικά ε, διαχειριζόντουσαν αυτά τα σχολεία καταφύγια. Οπότε όταν χρειάστηκε οι διαχειριστές των καταλημάτων, των καταφυγίων γίνανε δάσκαλοι. Βλέπετε επομένω το πώς ε, φροντίζουμε για την μακρόπνοη ανάπτυξη αλλά και τα κατεπήγοντα τα ανθρωπιστικά. Ε, επίσης πιστεύουμε ότι δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο για να παραμείνει εκεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ένα σημαντικό πρόβλημα είναι το, ότι είχε Ευρώπη τόσους Συρίους πρόσφυγες. Και αυτό σχετιζόταν με το πώς θα μπορούσαμε να παράσχουμε κάποιες σταθερές και ουσιαστικές υπηρεσίες βοήθειας. Επί πέντε χρόνια βοηθούμε για ολόκληρες γενιές Παλαιστινίων και τους δίνουμε απλώς εγγύηση, αλλά τη δυνατότητα να επιλέξουν να μείνουν εκεί. Και αυτά είναι γαλόνια που τα έχουμε, είναι δεδομένα. Και ξέρετε ότι οι φορολογούμενοι πληρώνουν με 9 φορές λιγότερα για να μας υποστηρίξουν όσον αφορά το να στηρίξουν αυτούς τους πρόσφυγες εκεί. Και θα δίνουν 7 με 9 φορές περισσότερα εάν αυτοί ερχόντουσαν εδώ. Βλέπετε επομένω πόσο ουσιαστική είναι η ωφέλεια από αυτή την ε, συνεργασία. Και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα που δίνουν όλοι οι δωρητές και οι Ευρωπαίοι φυσικά. Επίσης να σας τονίσω ότι το κόστος ανά μαθητή σας είπα ότι έχουν 500.000 μαθητές το κόστος ούτω ώστε να τους δώσουμε την παιδεία που χρειάζεται. Είναι 10% του κόστους που θα έπρεπε να καταβάλουν οι χώρες του ΟΣΑ στις χώρες τους για να εκπαιδεύσουν ένα παιδί. 10% δεν νομίζει για ένα μικρό Παλαιστίνιο και βέβαια οι βαθμοί που αποσπούν και οι επιδόσεις τους είναι φανταστικές. Το έλεγε και η Παγκόσμια Τράπεζα ότι η επιτυχία αυτή είναι δεδομένη παρά τις δυσκολίες και δεν το λέει αυτό η Παγκόσμια Τράπεζα γιατί μας δίνει λεφτά. Δεν μας δίνει. Είναι αντικειμενικό αυτό. Το λέει η Παγκόσμια Τράπεζα λοιπόν ότι στην Ιορδανία δεν δικαιώθηκε στη Γάζα ε, οι επιδόσεις των μαθητών είναι ίδιες ε, όπως και αλλού στα σχολεία. Να, και άλλο είναι επίτευγμα και γι' αυτό σας λέω ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας. Επίσης, το κόστος ανασθενεί στα νοσοκομεία μας. Είναι 1% του τι θα κατεβάλλεται στις χώρες του ΩΣΑ. 1 προς 5. Ε, πέντε φορές δηλαδή λιγότερο από ό,τι σε κάποιες χώρες μέσου και αποφασίσαμε φέτος, ακριβώς γιατί πέρσι είχαμε αυτό το χρηματοδοτικό πρόβλημα, να αναλάβουμε κάποιες εσωτερικές πρωτοβουλίες, ούτω ώστε να συγκρατήσουμε το κόστος. Γιατί θέλουμε όλοι οι εταίροι μας να μας βλέπουν ω αξιόπιστους όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων. Παραδείγματα. Πρώτον, κάποια εσωτερικά μέτρα ούτω ώστε να μειωθεί το έλλειμμα από 134 εκατομμύρια σε 74 εκατομμύρια. Μιλούμε για μια πάρα πολύ σταθή περιοχή και για να πετύχουμε αυτό χρειάστηκαν τρόμερες προσπάθειες. Δηλαδή, από το 2015 μέχρι το 2016 ο προπολογισμό δεν αυξήθηκε ούτε μία δεκάρα. Είμαστε ο μόνο διεθνή φορέα στη Μέση Ανατολή που είχαμε τη μηδενική αύξηση του προπολογισμού παρά το ότι οι ανάγκες γύρω τριγύρω εκεί αυξάνονται κάθετα. Βλέπετε πόσο σοβαροί είμαστε, ούτως ώστε να διαχειριστούμε καλά τη χρηματοδότηση. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που κάνουμε. Και φέτος κατά το πρώτο μας ε, εξάμεινο χαράξαμε μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική για να έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Τα είδη διατροφής, τα χρήματα, τα σχετικά κλπ. Θα τα πούμε. Οπότε βλέπετε τι γίνεται με εταίρου και τι γίνεται με δωρητέ. Όλα αυτά είναι σημαντικά και θα τα ξανασυζητήσουμε αυτή τη εβδομάδα για να δούμε ποια θα είναι η επόμενη φάση τη συνεργασία μα για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την υποστήριξη προ την Όνειρα και εμεί να αποδείξουμε ότι με αυτά τα μέτρα και μεταρρυθμίσει είμαστε σοβαροί και ότι θέλουμε η διεθνή κοινότητα να βρει μαζί μα λύσει και να μην ξανά έχουμε προβλήματα χρηματοδοτικά. Νέοι μηχανισμοί να υπάρξουν χρηματοδότηση. Ε, να ζητήσουμε λεφτά και τη Διεθνή Τράπεζα. Και γι' αυτό και θέλουμε και τα ευρωπαϊκά δεσμικά όργανα και οι ευρωπαίοι εταίροι να μα βοηθήσουν να ζητήσουμε λεφτά την Παγκόσμια Τράπεζα. Διότι έτσι θα υπάρξει περισσότερη σταθερότητα τη χρηματοδότησή μας στο μέλλον. Επίσης, στρεφόμαστε και στις χώρες του κόλπου, αλλά και στον Καναδά και αλλού. Επομένως και εμείς ε, έτσι θέλουμε να προχωρήσουν τα πράγματα. Τώρα κατακλείδη να σας πω κάποιες άλλες σκέψεις μου. Πρώτα, πρώτα σε με αυτό που είπα στην αρχή για την απουσία πολιτικού ορίζοντα, οράματος και λοιπά. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα βέβαια και θέλουμε ανθρωπιστική αρρωγή και ανάπτυξη. Έχω πιστεί από όλες μου τις αποστολές σε Συρία, σε Λίβανο, Γάζα, η Ορδανία, φυσικά και στη Δυτική Όχθη, έχω πιστεί λέγω ότι τίποτε δεν είναι πιο σημαντικό από το να ασχοληθεί επί του πολιτικού επέδου με το πρόβλημα η διεθνής κοινότητα. Και πολλές φορές με εκπλήσει το πόσο επιφυλακτική είναι σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, όχι μόνο στην Ευρώπη. Επιφυλακτικότητα σε σχέση με το τι μπορούν να πετύχουν στο μέτωπο της ειρήνευσης. Όμως, αυτή τη τακτικότητα μας οδήγησε στο σημείο που βρεθήκαμε σήμερα. Δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να συνεχίσει να, αντιμετωπίζει έτσι τη Μέση Ανατολία και να υφίσταται αυτές τις γνωστές συνέπειες χωρίς να αναζητείται κάποια εναλλακτική λύση. Έχουμε τις γαλλικέ πρωτοβουλίε. Έχουμε όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να γίνουν και θα πρέπει τελικά κάτι να κάνουμε για να υπάρξει φάρος ελπίδας. Γιατί αυτό χρειάζεται. Να ξαναδώσουμε ελπίδα, να ξαναδημιουργήσουμε εμπιστοσύνη, να μην υπάρχει αυτού του είδους όσμωση των διαφορετικών αφηγημάτων για τη Μέση Ανατολή. Να έχουμε μια σωστή διαδρομή που να στηθεί ε, από πλευρά τη πολιτική. Πολύ σημαντικό. Τώρα, ε, για την βοήθεια προ την Ούνρα, να σα πω. Είμαστε ευγνώμονε προ την Ευρώπη για τη βοήθειά σα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μα, για όσου δρούμε εκεί επί Και έχουμε, ξέρετε, χάσει πάρα πολλού συνεργάτε τα τελευταία χρόνια. Αυτοί που μα βοηθούσαν να υλοποιήσουμε τα όσα πρέπει. Νομίζω σας είχα πει ότι κατά την κρίση στη Γάζα χάσαμε 11 και τελικά άλλους 16 στη Συρία από τότε υπάρξει ο πόλεμος. 28 είναι δε οι αγνοούμενοι στην Συρία. Αλλά μιλάμε για την μεγαλύτερη κρίση που έχω υπόψη μου για οποιαδήποτε ανθρωπιστική πλατφόρμα και υπηρεσία. Να, πόσο θαραλέοι είναι οι συνεργάτες μας. Γι' αυτό και τους αξίζει κάθε τιμή και εκτίμηση. Και σας ευχαριστώ για την γενιοδορία σας προς την ούρα. Ιδίως τώρα. Ε, επίσης να σας πω όμως, γιατί αξίζει κανείς να βοηθάει. Πριν από ένα μήνα ήμουν στη Δαμασκό. Και... Εκεί ήμουνα μάρτυρας μιας φοβερής σκηνή. Πολλοί από εσά θα έχετε υπόψη σα τις εικόνες στη Γερμού κοντά στη Δαμασκό, μια γειτονιά όπου υπάρχει καταβλισμός της Δαμασκού ε, είναι πολύ γνωστός γιατί οικονομικά η περιοχή αυτή ήταν πολύ δυναμική πριν τον πόλεμο. 20.000 Παλαιστίνοι ζούσαν εκεί, τώρα είναι μια ερημιά. Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε μια από τις χειρότερες σκηνές καταστροφής μετά από πόλεμο, στο Γιαρούκο, ακριβώ εκεί. Λοιπόν, 20.000 όμω παραμένουν σε αυτό το καταβλισμό. Και όταν ήμουν στη Δαμασκό πριν από τέσσερι εβδομάδες, σε ένα από τα σχολεία έξω από τη Γιαρμούκ, εκεί συναντήθηκα με 120 μαθητές, οι οποίοι είχαν βγει την παραμονή από τον καταβλισμό Γιαρμούκ και ήταν στο σχολείο για να περάσουν εξετάσεις. Φανταστείτε λοιπόν τη σκηνή μέσα σε μια καταστραμμένη Συρία, μέσα σε μια καταστραμμένη γειτονιά της Δαμασκού είχατε 120 μαθητές, κορίτσια και αγόρια, Παλαιστίνους που βγήκαν από αυτή τη γειτονιά και πήγαν για να περάσουν τις εθνικές τους εξετάσεις. Και πέρσι ένας από αυτούς ήταν από τους καλύτερους μαθητές στη Συρία. Πώς το καταφέρνουν, πώς είναι δυνατόν να διατηρήσει κανείς ε, κάτι σαν μια εκπαιδευτική δομή μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα είναι πραγματικά θαύμα. Και όμως σύνολα το καταφέρνει αυτό εν μέρη με καινοτόμα μέσα προκειμένου να προσφέρει εκπαίδευση σε περιοχές όπου υπάρχει πόλεμος. Με υλικό για αυτούς τους μαθητές που δεν μπορούν να πάνε σε ένα σχολικό κτίριο προσφέρουμε με το κανάλι μας που έχουμε την έδρα στη Γάζα, υπάρχει τηλεόραση της Σούνρα. Οπότε μεταδίδονται προγράμματα που μπορούν να παρακολουθήσουν Παλαιστίνοι, αλλά όχι μόνο και Σύριοι και Ιρακινοί σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και το γεγονός ότι οι μαθητές αυτοί έχουν το θάρρος, το κουράγιο να βγουν από αυτές τις φρικτές σκηνές για να πάνε να περάσουν τις εξετάσεις τους, αυτό δείχνει πόσο σοβαρά σκέφτονται για την εκπαίδευσή τους και για το μέλλον τους οι άνθρωποι αυτοί, αυτά τα παιδιά. Τι προσδοκίες έχουν από τη ζωή τους. Και μια ακόμα ιστορία θα σας πω από τη Γάζα, όπου ένα νερό κορίτσι ήρθε στο πόντιου μαζί μου πριν από 1,5 μήνα είχε πάρει ένα πιστοποιητικό για τα επιτεύγματά της. Ονομάζεται AHEAD. Είναι 14 ετών. Καταστράφηκε το σπίτι της το 2014 με τη σύγκρουση στη Γάζα έμεινε για μήνες σε κόμμα και μόλις ξύπνησε από το κόμμα αυτό της είπαν ότι η μητέρα της και τα δυο της αδέρφια είχαν σκοτωθεί στην επίθεση και όμως είναι μια από τις καλύτερες μαθήτριές μας. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση παρά να σκεφτεί κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν ελπίδα μέσα από την απελπισία. Έχουμε τεράστια ελπίδα λοιπόν με αυτούς και έχουμε και τεράστια ευθύνη απέναντί τους με ανθρωπιστικά προγράμματα με εκπαίδευση και κυρίως με πολιτική δέσμευση όσον αφορά το Συριακό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λίτς, έχετε το λόγο. Α, προηγουμένως ο κύριος Βαϊράν, συγγνώμη. Α, θέλετε ο κύριος Λίτς, εντάξει, ο κύριος Λίτς τότε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, τόσο εντυπωσιακή παρουσίασή σας πέρσι υπήρξε μια κατάρρευση σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της παιδείας. Η παιδεία δεν είναι μόνο ένας πυλώνας ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά και ένας πυλώνας ασφάλειας. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και έχουμε ζητήσει να μάθουμε στην Κομισιόν, από την Κομισιόν να επενδύσει περισσότερο για την παιδεία. Ήταν πρωτοβουλία των σοσιαλδημοκρατών στο πρόγραμμα Εντούκα να, η πρότασή μας να δώσουμε περισσότερα κονδύλια για την παιδεία και να χρησιμοποιήσουμε και το Συριακό Ταμείο το οποίο έχει δημιουργηθεί στη διάσκεψη του Λονδίνου. Χαίρομαι λοιπόν που αναφέρεται και την ε, οικονομική βοήθεια της παγκόσμια Τράπεζα, αλλά έχετε πάρει κάποια χρήματα από του δωρητέ τη συνδιάσκεψης του Λονδίνου για τη Συρία και την γύρω περιοχή και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της διεθνού ανθρωπιστικής διάσκεψης για την παιδεία. Επίση, εμεί, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέμε κάθε φορά ότι δεν μας δίνουν την άδεια να πάμε στη Λωρίδα της Γάζας και εξαρτιόμαστε από τις εκθέσεις που μας δίνετε εσείς για τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται και τα χρήματα τα οποία παίρνετε για να δώσετε ελπίδα στον, στους ανθρώπους εκεί. Όταν λέτε 90% δεν έχουν βγει ποτέ από τη λεωρίδα της Γάζας, μου θυμίζει την κατάσταση που είχα ζήσει στην Ανατολική Γερμανία, που ήταν πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των ανθρώπων που δεν μπορούσαν να βγουν από τη χώρα τους. Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο για ένα νεαρό, ο οποίος ε, επέκρινε την ε, δίκηση της Χαμάς στη Γάζα, έκανε απεριαπίνα τον βάλαν στη φυλακή, δέχτηκε να μην μιλάει δημόσια, αλλά εξακολουθεί να αγωνίζεται για τα θέματα αυτά. Βλέπετε να υπάρχει μια μεγαλύτερη ομάδα νέων που είναι πολύ καλά μορφωμένοι, όπως αυτός ο νέος, και δεν βλέπουν το παραμικρό μέλλον. Μιλάτε για την ε, το ποσοστό των νέων που είναι άνεργοι. Υπάρχει μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που συζητούν για τα θέματα αυτά. Είναι μια κατάσταση που συζητείται για τη χαμάση μεταξύ μαθητών, καθηγητών. Αυτό θα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το έργο σας και περιμένω τις απαντήσεις σας. Ο κύριος Φρέντ. Φρόιντ, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κρέμπιλ για την τόσο συγκινητική σας και τόσο πλήρη και πληροφοριακή παρουσίαση που μας δείξατε, που μας δώσατε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας όταν λέτε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με αυτή την αντιπαράθεση από τον παρελθόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω όσο καιρό είμαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία δύο χρόνια και ως μέλος της αντιπροσωπείας με την Παλαιστίνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν από δύο μήνες ήμασταν στην περιοχή αυτή και πάλι όπως είπε και ο κύριος Λίτς δεν είχαμε το δικαίωμα να πάμε στην ε, Λόριδα της Γάζας, μόνο στη Δυτική Όχθη. Πάντα έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο μειονέκτημα ως αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να σταθώ σε κάποια από τα σχόλιά σας και θα ήθελα, να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Είπατε ότι υπάρχουν 500.000 φοιτητές στην ε, περιοχή αυτή. 500 αυτές χιλιάδες είναι σε όλους τους ε, βαθμούς της, σε όλα τα επίπεδα της παιδείας. Ξεκινάμε από δημοτικό και φτάνουμε μέχρι πανεπιστήμιο ή όχι. Και για τους διδάσκοντες. Χρησιμοποιείται ανθρώπους που είναι τοπικοί, είναι πολίτες εκεί της περιοχής ή φαίνεται περισσότερους δασκάλους από άλλα μέρη του κόσμου. Και τώρα για τον προϋπολογισμό με μηδενική αύξηση που αναφέρατε. Από τη μία πλευρά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά αυτά που κάνετε. Από την άλλη πλευρά σημαίνει αυτή η μηδενική αύξηση, ότι πρέπει να περικόψετε οι υπηρεσίες που είχατε τα προηγούμενα χρόνια. Και ένα ερώτημα που δεν είναι ακριβώς ε, συνδεόμενο με τη Γάζα και την Δυτική Όχθη, αλλά με τις εκατοντάδες χιλιάδες Συρίων, εκατομμύρια Συρίων προσφύγων. Κάτι που μας λένε πάντα είναι ότι δημιουργούμε μία γενιά παιδιών που θα, δεν θα έχουν την ευκαιρία να έχουν μόρφωση και επομένως θα αποτελέσουν μια ορολογιακή βόμβα για τα επόμενα χρόνια. Τι είδους υπηρεσίες <clears throat> μπορείτε εσείς να προσφέρετε, αν μπορείτε να προσφέρετε, για τα παιδιά των Συρίων προσφύγων και κατά πόσο γίνεται κάτι για τα θέματα αυτά. Γιατί ξέρουμε ότι είναι ευρέως κατανεμημένη στην Μέση Ανατολή σε πολλά μέρη. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το έργο σας ως επικεφαλής Σούντρα. Παρακαλώ για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα για τον κύριο Λίτς. Όσον αφορά την εκπαίδευση, πράγματι είναι αναγκαίο να επιμείνουμε όλο και περισσότερο σε αυτό. Το ομολογώ δημόσιο ότι αυτό το αντιλήφθηκα από τότε που συμμετέχω στην Ούνρα. 20 χρόνια ήμουνα στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού σε περιοχές με συγκρούσεις. Πρέπει να ομολογήσω ότι όπως και πολλοί έχω Πιστεί ότι όταν ξεκινάει ένας πόλεμος σκεφτόμαστε πώς θα δώσουμε τρόφιμα στον κόσμο, ιατρική περίθαλψη, πώς θα τους προστατεύσουμε. Το θέμα της εκπαίδευσης όμως πάντα σκεφτόμαστε ότι πρέπει να το αφήσουμε για αργότερα, για καλύτερους καιρούς. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια, γιατί στην πραγματικότητα κάτι διαφορετικό θέλει ο κόσμος στις περιοχές αυτές που βρίσκονται σε σύγκρουση. Θυμάμαι από εκθέσεις της Επιτροπής όπου μιλούσαμε με κοινότητες σε έξι διαφορετικές περιοχές όπου υπήρχε πόλεμος, μεταξύ άλλων και στο Αφγανιστάν. Ρωτούσαμε λοιπόν τον κόσμο ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες, προκλήσεις που αντιμετώπιζαν, ποιες θα ήταν οι προτερότητε τους. Και στην έκθεση που διάβασα για το Αφγανιστάν, όταν ρωτήθηκε ο κόσμος στο Αφγανιστάν, απάντησε ότι η πρώτη τους ανησυχία βέβαια ήταν το θέμα της ασφάλειας, δεν μας εκπλήσει. Το δεύτερο όμως που έβαλαν στον κατάλογο στη σειρά ήταν η εκπαίδευση. Τότε δεν ασχολιόμασταν τόσο πολύ με την εκπαίδευση και μου είχε κάνει εντύπωση αυτή η απάντηση. Μπορεί να ήμασταν αφελείς ή να μην είχα εμπειρία. Πάντως ήταν ξεκάθαρο τελικά ότι όταν ρωτάς τον κόσμο αυτοί ξέρουν ότι όσο και αν κρατήσει ένας πόλεμος κάποια στιγμή θα τελειώσει. Και αν δεν έχουν γίνει επενδύσεις στην εκπαίδευση τα προβλήματα θα είναι μεγάλα μετά. Οπότε συλλογικά όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε τη σημασία που έχει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και κυρίως να διατηρήσουμε τις δομές της εκπαίδευσης και μέσα σε ένα πόλεμο. Και θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ένα από τα πράγματα που με έχουν εκπλήξει όσον αφορά τις ικανότητες της Σούντρα είναι ότι αυτό μπορεί να το κάνει, να διατηρήσει δηλαδή τις εκπαιδευτικές δομές ακόμα και σε ένα σταθές περιβάλλον. Στη Συρία για παράδειγμα πρόσφατα είδα ότι ένα σχολείο που επισκέφτηκα πριν από ένα χρόνο, που καταστράφηκε από ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο. Ήταν κενό το σχολείο. Τώρα η Ούνρα το ξαναχτίζει σε μια από τις καταστραμμένες περιοχές ε, της Συρίας. Είναι ένα δείγμα δηλαδή ότι δεν παρετούμαστε, δεν παρετούμαστε από την εκπαίδευση και δεν πρέπει να μιλάμε θεωρητικά για την εκπαίδευση. Δεν αρκεί να μοιράζουμε υλικό <coughs> εκπαιδευτικό, δεν αρκεί να συναντιόμαστε σε διεθνές επίπεδο, σε σεμινέρι. Όχι, επί τόπου πρέπει να προσφέρουμε την εκπαίδευση και η UNRWA το κάνει αυτό. Και θα επανέλθω και αργότερα. Οπότε ναι, πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασία να υπογραμμίσουμε το θέμα της εκπαίδευσης. Είναι μια επένδυση που κάνουμε για το μέλλον και για τη μελλοντική σταθερότητα. Σκεφτείτε στην περίπτωση των Παλαιστινίων. Έχετε αυτή την τραγική ηρωνία. Πρόκειται για μια κοινότητα που συνεχίζει να αναπτύσσεται εξαιτία τη θέληση των ίδιων των Παλαιστινίων. Γιατί δεν τους προσφέρουμε εμείς την εκπαίδευση, είναι εκείνοι που φροντίζουν, χωρίς κράτος. Πολλέ χώρες έχουν αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα, αλλά δεν διαθέτουν το ανθρώπινο δυναμικό για να αναπτυχθούν. Ενώ οι Παλαιστίνοι που δεν έχουν κράτο έχουν το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο υποστηρίζει την εκπαίδευση. Αυτό πρέπει λοιπόν να το έχουμε υπόψη μας. Είπατε τι έγινε με τη διάσκεψη του Λονδίνου για την οικονομική στήριξη. Ένα από τα πράγματα που ζητήσαμε στο Λονδίνο είχε να κάνει με ε, χρήματα προς την Ούρα. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα για επιπλέον χρήματα. Όσον αφορά την επίγουσα ανάγκη δηλαδή, μπορεί να έχουμε περισσότερα χρήματα. Πάντως συνολικά δεν έχει αλλάξει κάτι. Για τους λόγους που και εσείς αναφέρετε, καταγράφουμε τι προσφέρουμε επιτόπου και ότι επιπλέον χρήματα βρεθούν στο δρόμο μας θα χρησιμοποιηθούν επίσης αμέσως. Είμαι ευγνώμων πάντως για το γεγονός ότι ακόμα και στο ευρωπαϊκό επίπεδο είχαμε κάποια στήριξη όταν θέσαμε το θέμα των Παλαιστινίων προσφύγων στη διάσκεψη αυτή του Λονδίνου και ο Επίτροπος Χάν και άλλοι ε, το σημείωσαν. Ο κίνδυνος είναι ότι θα τους ξεχάσουμε τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι σημαντικό γιατί όντως υποστηρίζει τους πρόσφυγες γενικά, αλλά πιο συγκεκριμένα την εκπαίδευσή τους. Το πάνελ ήταν πολύ καλό η Ειρήνα Μπόκοβα, ο Μπράουν, Κίλαρ και άλλοι ήταν παρόντες και ήταν σημαντικό που συζητήσαμε. Είχαμε πολύ καλή συζήτηση με τον Γκόρντον Μπράουν για το θέμα της εκπαίδευσης. Στη συνάντησή μου είπε ως ειδικό απεσταλμένο για την ε, παγκόσμια εκπαίδευση η UNRWA είναι ο οργανισμός που προσφέρει περισσότερο να τον κόσμο. Υπάρχει βέβαια και η UNESCO, αλλά μέσα στα σχολεία, απευθείας δηλαδή εκπαίδευση με δασκάλους, είναι η UNRWA, ο μεγαλύτερος οργανισμός και πρέπει να διατηρηθεί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα για το σχόλιο σα όσον αφορά επίσκεψη στη Γάζα. Πράγματι, πολύ σημαντικό. Τίποτα δεν αντικαθιστά μια επίσκεψη επιτόπου. Και θα σα δώσω παράδειγμα Πολλές επισκέψεις από τους διπλωμάτες, υπουργούς κτλ. έχουν γίνει στη Δυτική Όχθη, στη Γάζα που συναντιόνται με τους τοπικούς βουλευτές. Να ξέρετε ότι και για την Ούνρα είναι πάρα πολύ σημαντικό οι δάσκαλοι μας εκεί και ο κόσμος της Ούνρα να συναντηθούν μαζί σας, να κοιταχτείτε στα μάτια, να σας πούνε τι κάνουν στα σχολεία ποιες είναι οι προτεραιότητες στα σχολεία, στις, ε, τι υπηρεσίε προσφέρουν για τους ηλικιωμένους κτλ. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο να μας πούνε, να μπορέσουν να μας πούνε τι περιμένουν από μας και να μην υπάρξει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο. Η συνάντηση λοιπόν με τα σχολικά κοινοβούλια είναι τεράστια σημασίας. Ήδη από φέτος το καλοκαίρι θα αρχίσουμε με εκπροσώπους από όλα τα σχολικά κοινοβούλια και θα ξεκινήσουμε νέες πρωτοβουλίες υπέρ της νεολαίας. Και αν πάτε και τους επισκεφθείτε ή αν κάποιοι από αυτούς έρθουν εδώ και σας συναντήσουν στις Βρυξέλλες, θα ήταν πολύτιμο. Ο πρόεδρος Σούλτς ξέρω ότι έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για να αρχίσουν και πάλι επισκέψεις στην Γάζα. Είναι ένα σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει. Με ρωτήσατε, αν κατάλαβα καλά την τελευταία σας ερώτηση, κατά πόσο γίνονται συζητήσεις ανάμεσα στους μαθητές, στο προσωπικό για την κατάσταση που επικρατεί μέσα στη Γάζα. Επ' αυτού το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι καθημερινά αναλύει ο κόσμος εκεί την κατάσταση που τον αφορά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα είναι επικριτική όσον αφορά τις συνέπειες όπως τις αντιλαμβάνονται από την κατοχή του Ισραήλ. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα είναι επικριτική και απέναντι στους αυτούς τους ε, συχνά όσον αφορά την έλλειψη ενότητας στην Παλαιστίνη ότι είναι κατακαιρματισμένοι ήδη οι Παλαιστίνοι, αλλά είναι επικριτική και απέναντι στη διεθνή κοινότητα. Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, για παράδειγμα, θεωρούν ότι έχει προδώσει τις ελπίδες τους, τις προσδοκίες τους. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Αλλά αυτό που πρέπει να θυμόμαστε επίσης είναι ότι στα σχολιά μας αυτό που προσπαθούμε να διδάξουμε είναι και πράγματα τα οποία είναι συμβατά με τις αξίες μας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για παράδειγμα, έχουμε ένα τέτοιο μάθημα που επικεντρώνεται ε, πολύ στο να ε, μαθαίνουμε τι συμβαίνει αλλού, στην Ευρώπη, στην Αφρική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να συνδυτοποιήσουν οι νέοι που ακριβώς βρίσκονται και τι συμβαίνει γύρω τους. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι συζητούν για την ε, δικιά τους κατάσταση και είναι επικριτικοί και απέναντι στους εαυτούς τους, όπως και απέναντι στους γειτονές τους και τη διεθνή κοινότητα. Κάτι άλλο τώρα για το σχόλιο σας όσον αφορά την Ευρώπη, κατά πόσο θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Στο τέλος των παρατηρήσεων μου κάτι σας είπα σχετικά, αλλά πιο συγκεκριμένα για τους 500.000 μαθητές. Πάνε από εντάξει 1 έως 9. Και μερικές φορές πάνε και στην δέκατη τάξη. Δεν μπορούμε να τους πάμε πιο πέρα, ούτε προσφέρουμε όλα τα μαθήματα στο επίπεδο 10. Δεν είναι αυτό εφικτό. Τεχνικά θα μπορούσαμε και για μένα θα ήταν σημαντικό να επεκτείνω τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της Ούνρα ακόμα περισσότερο. Βέβαια θα μου πείτε και γιατί όχι ενδέκατος χρόνος και δωδέκατος. Αλλά αυτό που έχουμε είναι το σχολικό μας πρόγραμμα που είναι συμβατό με το εθνικό εκεί όπου διδάσκουμε. Αν είναι στην Ιορδανία, τότε το σχολικό πρόγραμμα είναι όπως το Ιορδανικό σχολικό πρόγραμμα, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να πάνε στο πανεπιστήμιο ενδεχομένω στη χώρα στην οποία έχουν κάνει και το σχολείο τους. Οι δάσκαλοι και το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι 20.000 δηλαδή της UNRWA που δουλεύουν στην εκπαίδευση είναι όλοι Παλαιστίνοι με ελάχιστε εξαιρέσει. Ο διευθυντή του εκπαιδευτικού μα προγράμματο ή κάποιοι στην έδρα μα. Κατά τα άλλα, είναι όλοι Παλαιστίνοι. Όπως είπα και νωρίτερα, το 98% του προσωπικού της Ούνουρα είναι Παλαιστίνοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια τεράστια αξία για την περιοχή. Οι δυνατότητες, οι ικανότητες, όλα αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε, πρόκειται για συναδέρφους με τεράστια εμπειρία. Στην Ρούρου είναι 30.000 το προσωπικό, με 40.000 χρόνια εμπειρία. Δύσκολα μπορεί κανείς να βρει καλύτερα για τον προπολογισμό που δεν αυξάνεται, εμείς περιορίζουμε τις δαπάνες. Πήραμε κάποια σκληρά μέτρα πέρυσι. Αυξήσαμε το μέσο όρο του αριθμού μαθητών ανατάξει. Έχει βέβαια αυτό κάποιες επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης, το ξέρουμε. Από 38,5 πήγαμε στους 39,5 μαθητές ανατάξει. Δηλαδή κάπου μπορεί να έχουμε 50 μαθητές ανατάξει. Αλλού βέβαια λιγότερα. Ε, η πίεση είναι μεγάλη, είναι ένα δύσκολο ζήτημα αυτό. Και ένα από τα μέτρα που πήραμε φέτος θα, θα αναλυθούν και θα θεωρηθούν ίσως ως μείωση υπηρεσιών. Έχουμε κάνει μια αλλαγή από τροφιμική βοήθεια με πακέτα τροφίμων σε ε, χρήματα ή σε κουπόνια για τρόφιμα. Γιατί το θέμα της διανομής τροφίμων είναι κατά κάποιο τρόπο μια υπενθύμηση ότι είναι πρόσφυγες. Αλλάξαμε προ ένα σύστημα που είναι πιο αξιοπρεπέ, δίνει τη δυνατότητα στου ανθρώπου να διαλέγουν, αντί να παίρνουν πάντα τα ίδια τρόφιμα, να διαλέγουν αυτοί τι τρόφιμα θέλουν να αγοράσουν στι τοπικέ αγορέ. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά δεν πηγαίνουν στο εξωτερικό για να αγοραστούν τα τρόφιμα και να έρθουν στην ε, Παλαιστίνη, αλλά αγοράζονται στην τοπική αγορά, το οποίο έχει και εκεί θετικό αντίκτυπο. Καταλαβαίνω όμως γιατί οι ορισμένοι πρόσφυγες λένε αυτό που συμβαίνει ότι παίρνω 120 δολάρια το χρόνο αυτή τη στιγμή, αλλά να αλλάξει η οικονομική κατάσταση θα παραμείνει σταθερό το, ε, η αγοραστική δύναμη που μου δίνουν αυτά τα, χρήματα. Γι' αυτό υπάρχει η αντίληψη μερικές φορές ότι περιορίζονται οι υπηρεσίες. Κάτι ακόμα που πρέπει να σας υπενθυμίσω. Αν η πατιαρμοστία για τους πρόσφυγες μειώνει τον προϋπολογισμό της ένα χρόνο, έχει να αντιμετωπίσει πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο δεν ξέρει κάποιος αν η απόφαση της μείωσης τους ε, θίγει άμεσα. Αλλά εμείς το ξέρουμε στην περίπτωση της Ούρα, γιατί είμαστε το βαρόμετρο για την τοπική κοινότητα των Παλαιστινίων. Αν ξέρουν λοιπόν οι Παλαιστινοί ότι αλλάζει ο προγραμματισμός στην Ούρα, αν μιλήσουμε για μεταρρύθμιση, φοβούνται ότι αυτό είναι απλώς καλοπισμός των περικοπών. Είναι φυσιολογικό αυτό, έχουν περάσει τόσο μεγάλες απογοητεύσεις, τόσες ε, προδοσίες όπως τις αντιλαμβάνονται για γενιές που είναι καχύποπτοι. Μίλησατε για τους ε, Σύριους και τα παιδιά τα οποία τη γενιά αυτή που δεν έχει εκπαιδευτεί και τις υπηρεσίες μπορεί να δώσει ουρά. Είναι τεράστιο το θέμα αυτό. Ένα τεράστιο πρόβλημα που έχετε πια μπροστά σας. Είναι η δεύτερη σε μέγεθος πια κοινότητα σε μέγεθος προσφύγων στη Μέση Ανατολή που ζει δίπλα-δίπλα με τους Παλαιστινίους. Είναι περίπου το ίδιο μέγεθος 5 εκατομμύρια και είναι άτομα τα οποία δεν έχουν την ίδια σταθερή πρόσφυ, πρόσβαση στην παιδεία όπως η Παλαιστίνη. Για πολλούς λόγους που καταλαβαίνετε η ώρα δεν μπορεί να δώσει υπηρεσίες ε, παιδείας στους Σύριους πρόσφυγες αυτό, γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα της ε, είπα της αρμοστίας για τους πρόσφυγες. Αλλά το είπα αυτό και στην ανθρωπιστική διάσκεψη ότι ο κόσμος μπορεί να χρησιμοποιήσει καλύτερα την εμπειρογνωμοσύνη και τη γνώση της Ούνρα για να βοηθήσει τις μακροχρόνια προσφυγικές κοινότητες. Έχουμε κάνει σφάλματα, αλλά έχουμε πετύχει και πράγματα. Σίγουρα έχουμε αποκομίσει κάποια εμπειρία. Αν είχαμε τα μέσα <clears throat> που ίσα ίσα καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα με τα χρήματα που έχουμε. Αν είχαμε τη δυνατότητα και υπήρχε η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας για να βοηθήσουμε άλλους φορείς που ασχολούνται με τους Σύριους πρόσφυγες εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θα υπήρχαν Παλαιστίνοι ε, διδάσκοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να εμπλακούν σε αυτά σε αυτήν την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Αλλά αυτό φυσικά αν έχουμε καλύψει τι δικέ μα εκπαιδευτικέ ανάγκε. Τελευταία παρατήρηση, γιατί μίλησατε για την ευρωπαϊκή παρουσία και τον ευρωπαϊκό ρόλο. Σε όλε τι επισκέψει μου στι ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε του τελευταίους μήνε είδα να υπάρχει μια πραγματική πρόκληση. Υπάρχει μια δοκιμασία καταρχήν Εγώ έρχομαι από μια χώρα που δεν είναι βέβαια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πολλοί από τους ε, συμπολίτες μου μερικές φορές νιώθουν ότι δεν ζουν στην Ευρώπη. Ως Ευρωπαίοι πάντως έχουμε ενώπιον μας μια δοκιμασία στις χώρες μας. Πολλοί από εσά το βλέπετε πηγαίνω σε συναντήσεις, σε συνδιασκέψεις. Βλέπω πόσο έντονα συναισθήματα δημιουργούνται στους πολίτες Ευρώπης. Κάποιες φορές δικαιολογημένα για την έλευση των μεταναστών και των προσφύγων, εδώ η Ευρώπη, η οποία υποστηρίζει το σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, προσφυγικού δικαίου, όταν αναφέρεται σε χώρες σε άλλα μέρη του κόσμου, ίσως πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να τακτοποιήσει και τα, του οίκου της και να καταλάβει ότι η παγκοσμιότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι απτή και στην ίδια Ευρώπη και θα πρέπει να τηρούμε τις αξίες αυτές που βρίσκονται στις συνθήκες μας. Εγώ δούλεψα για την, για την Επιτροπή του Ερθρού Σταυρού μετά από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου. Και θυμάμαι αυτούς που είπαν και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη ότι θα έπρεπε να επικαιροποιηθεί η σύμβαση της Γενέβης. Γιατί κανείς από αυτούς που διαπραγματεύτηκαν το 1949 τη Σύμβαση Γενέβης είχε προβλέψει κινήσεις όπως αυτές της Αλκάιντα ή άλλα φαινόμενα. Μπορεί να είναι αλήθεια αλλά αυτοί που έκαναν τις διαπραγματεύσεις το 1949 χρειαζόταν κάποια άλλη έμπνευση από την παραφροσύνη και την καταστροφή που έχει επιβάλει η ανθρωπότητα στον εαυτό της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η δήλωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Σύμβαση της Γενέβης, η Σύμβαση των, για τους πρόσφυγες είναι αποκοίημα της καταστροφής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας σοβαρά. Εάν δεν λάβουμε λοιπόν υπόψη αυτά που προήλθαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αμφισβητούμε αυτές τις ε, συμβάσεις και αυτούς τους κανόνες και τη σημασία τους για τη συνολική ασφάλεια και αξιοπρέπεια των ανθρώπων, τότε δημιουργούμε προβλήματα πολύ μεγάλα. Θα κάνω ένα, μια παρομοίωση του Λίβανου με την, με την ε, Ελβετία. Ο Λίβανος έχει το μισό πληθυσμό της Ελβετίας. Δηλαδή εμείς αναλογικά με το Λίβανο, θα έπρεπε να είχαμε 3 εκατομμύρια Αυστριακούς. Όπως ο Λίβανος έχει πάρει 1,5 εκατομμύρια, ε, Σύριους. Φανταστείτε την, ε, την Ελβετία να έχει πάρει 3 εκατομμύρια ε, Αυστριακούς όταν υπάρχει μια ιστερική συζήτηση όταν τίθεται το θέμα να υποδεχτούμε χιλιάδες, όχι εκατομμύρια ανθρώπους αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη δεν θα μπορέσουν να πάψουν να συμβαίνουν, αν δεν καταλάβουμε πραγματικά τις πηγές αστάθειας που οδηγεί στη μετακίνηση τόσων ανθρώπων. 25 χρόνια που εργάζομαι σε εμπόλεμες περιοχές, δεν έχω δει ποτέ ένα εκτοπισμένο ή ένα πρόσφυγα που θέλει να είναι εκτοπισμένος ή πρόσφυγας. Ποτέ δεν είδα κάποιον ο οποίος θέλει να παραμείνει πρόσφυγας. Και ποτέ δεν είδα κανένα ο οποίος θέλει να είναι πρόσφυγας μακριά από, τι από τις αιστείες του από το σπίτι του και όχι κοντά στο σπίτι του. Είναι δική μας ευθύνη να εξασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές διαδικασίες που ακολουθούμε είναι ουσιαστικές και δεν μιλάω για την διαχείριση κρίσεων και αντιπαραθέσεων. Η διαχείριση συγκρούσεων μας έχει φέρει εδώ που είμαστε. Μπορείτε να διαχειριστείτε αυτέ τι συγκρούσει για 50 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχετε δώσει μια λύση στου ανθρώπου, δεν του έχετε ξαναδώσει την αξιοπρέπεια του. Χρειαζόμαστε επίλυση συγκρούσεων. Να τελειώνουν κάποια στιγμή όχι απλώ να τι διαχειρίζουμε. Η Ούγγρα μπορεί να συνεχίσει άλλα 65 χρόνια, αλλά αυτό δεν είναι η απόδοση αξιοπρέπεια στου Παλαιστινίου ούτε η εξασφάλιση της σταθερότητα και της ειρήνη για όλους τους άλλου. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Βαύριν, ο τελευταίος μας ομιλητής. Είναι η τέταρτη φορά που η ευγένειά σας είναι η αιτία που μου δίνετε το λόγο. Να ευχαριστήσουμε τον εκπρόσωπο της Σούντρα για την εισήγησή του. Εγώ θα κάνω όπως ο Έλμαρ. Μας τα είπε στα γερμανικά και τώρα να φορέσει τα ακουστικά σας γιατί εγώ θα ολοκληρώσω τη συνάντηση μιλώντας στα φιλανδικά. Κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Βαρίνεν, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του κυρίου Κρένμπουλ. Αυτό που ήλθε στο ενδιαφέρον μου είναι το πώς ο πόλεμος στην Συρία επιδρά στο έργο της Ούνρα και το πώς βοηθά τους Παλαιστινίους η Ούνρα, κάτι το οποίο είναι παράγον σταθερότητας για την Μέση Ανατολία. Βλέπουμε δηλαδή πως ευρύτερες είναι οι συνέπειες του έργου της ε, UNRWA που βοηθά τόσο πολύ τα παιδιά και τους νέους. Εξεπλάγει πάντως από τον αριθμό των θεμάτων, εν μέσω των συνεργατών της ε, Ούνρα. Φυσικά και πρέπει να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για τους συνεργάτες της ε, UNRWA. Η Επιτροπή Ανάπτυξης δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Ακριβώς, όπως είπαμε όμως, ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να γινουν χερι χέρι-χέρι. Και εγώ και ο κύριος Σαλόμ έχουμε ασχοληθεί με μια γνωμοδότηση σε σχέση με την συνάντηση κορυφής για την ανθρωπιστική βοήθεια. Εστιάσαμε την προσοχή μας στην Επιτροπή μας στο πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά. Αυτά είναι προβλήματα πάγια και στις μακρόχρονες κρίσεις και στις πιο σύντομες. Το προσωπικό της Σούνερα έχει συνεργαστεί και με τη δική μας Επιτροπή. Έχουμε ασχοληθεί και με εκείνες τις ημερίδες ανάπτυξης. Στο πάνε είχαμε και την Πρωθυπουργό της ε, Αυστραλίας. που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις ανθρωπιστικές προσπάθειες. Ελπίζουμε αυτό το πάνελ τελικά να πετύχει στην αποστολή του και να συνεχιστεί η καλή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής μας, με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και της ούνερα Θερμές ευχαριστίες για τα όσα μας είπατε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κράινμπιουρ και, και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε του χρόνου να ακούσουμε περισσότερα για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Κλείνω τη συνεδρία αρχίζουμε αύριο σε 9.